Όπως βλέπετε, βέβαια, η πολιτική μηδενικών, μηδενικής αύξηση στο προσωπικό είναι αρκετά δύσκολη γιατί υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα έχουμε περισσότερο προσωπικό στη διάθεσή μας. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε να, να κατατάξουμε τον κόσμο που έχουμε από τη μία γενική διεύθυνση στην άλλη ε, εκεί όπου θα χρειαστεί να δουλέψουν όλοι πολύ σκληρά ε, πράγμα που σημαίνει με, ότι θα πρέπει να ασκήσουμε μια πολύ ευφυή πολιτική προσωπικού στην Κομισιόν. Και για να κάνουμε τέτοιο είδους πολιτική πρέπει να έχουμε πολύ καλή ενημέρωση. Στην διαφάνεια βλέπετε ποια είναι η σημερινή στελέχωση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Βλέπετε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το μεγαλύτερο θεσμικό όργανο, αλλά ταυτόχρονα βλέπετε αυξήσεις προσωπικού στα θεσμικά όργανα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 11 ετών. Θα παρατηρήσετε ότι η αύξηση του προσωπικού στην Κομισιόν ήταν η μικρότερη. Τώρα, για την ε, Κομισιόν, σε αυτόν τον ε, πίνακα, εδώ θα δείτε ποιος είναι ο διαχωρισμός ε, του προσωπικού μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά ολόκληρη, όλα τα θεσμικά όργανα, έχουμε συνολικά γύρω στις 40.000 θέσεις. Και σε αυτές πρέπει να προσθεθούν 10.000 άνθρωποι που εργάζονται ως, με προσωρινές συμβάσεις. Αν έρθουμε τώρα και στραφούμε στην Κομισιόν. Αυτή είναι η κατάσταση που βλέπετε στην εικόνα. Έχουμε 35.500 ε, υπαλλήλους θα δείτε πως έχουμε ε, υπαλλήλου ε, αορίστου χρόνου περισσότερο και προσωρινούς, ε, προσωρινές συμβάσεις και μετά έχουμε και τοπικό προσωπικό που είναι λιγότερο από το 10% και περισσότεροι εξ αυτών εργάζονται στα γραφεία μας σε τρίτες χώρες. Επιπλέον, όταν μιλάμε για το screening, για τον έλεγχο, δεν περιοριζόμαστε μόνο στο προσωπικό εξετάζουμε και τους ανθρώπους που προσφέρουν υπηρεσίες στην Κομισιόν επί τη βάση διαφόρων ειδών συμβάσεων ή επί τη βάση ε, χορηγιών. Μιλάμε για τους ερευνητές που δουλεύουν στα διάφορα ερευνητικά μας ιδρύματα και για τους εμπειρογνώμονες. Ακόμα δηλαδή 5.500 άνθρωποι. Στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε πώς μετατρέψαμε τη διαδικασία ελέγχου στην Κομισιόν. Όπως ξέρετε, είχε γίνει μόνο μία μελέτη το 1991 σχετικά. Ε, τότε εκφράστηκαν πολλές επιφυλάξεις σε σχέση με τη μέθοδο ελέγχου και γιατί. Γιατί δουλέψαμε με στοιχεία τα οποία συλλέξαμε από κάτω, δηλαδή από τις γενικές διευθύνσεις. Τώρα αλλάξαμε στάση και εργαζόμαστε με εργαλεία πληροφορικής και με τις πληροφορίες που έχουμε στην Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, στη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού και η ανάλυση γίνεται από εμά και μόνο επικυρώνεται από τις Γενικές Διευθύνσεις. Έχουμε πολύ συγκεκριμένους αριθμούς περιγραφές των θέσεων και μπορούμε να είμαστε ε, σίγουροι ότι τα στοιχεία, που, τα αριθμητικά που σας δίνουμε είναι σωστά. Σε σχέση με επενδύσεις που κάναμε, ε, για την προετοιμασία αυτού του ελέγχου. Μόνο το 5% εργάζεται κατά τη διάρκεια 12 μηνών για να προβεί σε αυτή την ανάλυση και νομίζω πως είναι μια αξιόλογη επένδυση η οποία μας δίνει μια σταθερή βάση για να λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις. Όταν συνάντησα κάποιους από εσά, συζητήσαμε όχι μόνο μεθοδολογία, αλλά και τις κατηγορίες του screening. Δηλαδή, να δούμε πόσο υπολογίζουμε, ποιοι ανήκουν στο επιχειρησιακό τμήμα, ποιοι θεωρείται ότι δουλεύουν για ουδέτερες υπηρεσίες και ποιοι ως βοηθητικό προσωπικό. Μιλάμε για τις διάφορες μονάδες. Όταν μιλάμε για το βοηθητικό προσωπικό, μιλάμε για τις διάφορες μονάδες και το προσωπικό που δουλεύει στην διοικητική στήριξη και στο συντονισμό. Στις ουδέτερες μονάδες μιλάμε για οικονομικό έλεγχο ε, γλωσσικές υπηρεσίες και καταπολέμηση των απατών να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό. Αν δείτε το χάρτη, θα δείτε πως είμαστε πάρα πολύ αυστηροί ε, όσον αφορά το πώς αξιολογούμε την περιγραφή των θέσεων των υπαλλήλων μας. Γιατί αν δούμε την διοικητική στήριξη, θα δούμε ότι η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού θεωρείται τέτοια υπηρεσία το 85% αυτής της υπηρεσίας και θέλω να θέσω την ερώτηση αυτή. Σε ποια χώρα θεωρείται βοηθητική υπηρεσία το Υπουργείο Οικονομικών Νομίζω σε καμία. Γι' αυτό το λέω για να σας δείξω ότι είναι το ότι είμαστε πολύ αυστηροί και ο Γιάννος Λεβαντόφσκι ε, λέει το ίδιο που είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με τις, ε, τον προπολογισμό. Έχουμε επίσης ε, τους εκπροσώπους μας, τους εκπροσώπους μας στα κράτη-μέλη που πρέπει να ενημερώνουν για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ σημαντικές θέσεις. Επίσης και μπορώ να προχωρήσω με τέτοιου είδους διευθύνσεις γιατί δεν μας δίνουν μόνο λύσεις στην πληροφορική αλλά είναι πολύ σημαντική για το την ε, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική διαμεθοριακή συνεργασία και ούτω καθεξής. Όταν μιλάμε για ουδέτερες ε, λειτουργίες, Μιλάμε και για τις γλωσσικές υπηρεσίες που χρειαζόμαστε για τη μετάφραση. Οι υπόλοιποι υπάλληλοι είναι στον επιχειρησιακό τομέα. Πώς έχει κατάσταση λοιπόν μετά τον τελευταίο αυτό έλεγχο. Θα δείτε εδώ ότι μετά από αυτό τον περιοριστικ... την περιοριστικού τύπου κατηγοριοποίηση θα δούμε ότι οι διοικητικές και οι συντονιστικές λειτουργίες καλύπτουν το 29,5% και ότι υπάρχει μια σταθερή μείωση του συνόλου του διοικητικού κομματιού και των σχετικών δαπανών στην Κομισιόν. Το μεγαλύτερο τμήμα των υπαλλήλων εργάζεται στους επιχειρησιακούς τομείς. Διαφορετικά, αν αφαιρέσουμε αυτό το προσωπικό που υπηρετεί άλλα θεσμικά όργανα, γιατί τους προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ε, όσον αφορά τις πληρωμές, οι λύσεις ε, πληροφορικής ή στις κοινέ δημοσιεύσεις και άλλες ε, υπηρεσίες όπου η Κομισιόν προσφέρει τις υπηρεσίες γιατί προσπαθούμε να κάνουμε οικονομίες κλίμακας όσον αφορά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και για να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες από πλευράς Κομισιόν αν αφαιρέσουμε αυτούς όλους και τους σταζιέρ θα ήμασταν στο 26,7%. Και πρέπει να προσθέσω ότι πρέπει να δούμε αυτό, αυτά τα στοιχεία από την προοπτική του τι είδους θεσμικά, θεσμικά όργανα είμαστε. Έχουμε γλωσσικές πιέσεις. Ξέρετε ότι βρισκόμαστε σε 170 ε, μέρη, διαφορετικές τοποθεσίες και επίσης πρέπει να μιλήσουμε και για υπηρεσίες που δεν είναι πολύ συνηθισμένες για άλλα διοικητικά όργανα. Επισκέφθηκα το ΙΣ πριν από δύο εβδομάδες και θα σας εκπλήξει το ότι και εκεί είμαστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση των οδικών, ε, του οδικού δικτύου, για την πυρηνική ασφάλεια και έχουμε ειδικευμένο προσωπικό που φροντίζει τη σημαντική αυτή ερευνητική μονάδα. Και όλα αυτά φυσικά κοστίζουν. Τώρα, τι κάνουμε με αυτά τα αποτελέσματα. Πώς θα πρέπει να τα ερμηνεύσουμε. Καταρχήν χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες ώστε να μειώσουμε τις διοικητικές δαπάνες όσο γίνεται με συγκεκριμένα όρια και κατόφλια. Αυτό είναι, σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να έχουν πάνω από 12% διοικητικές δαπάνες. Και αν δεν το καταφέρουν αυτό, πιέζουμε πολύ για να ανταποκριθούν σε αυτό το κριτήριο και άρα να μειωθούν οι διοικητικές δαπάνες όσο γίνεται περισσότερο. Επίσης εξετάζουμε ad hoc screening για τη Eurostat γιατί εκείνοι μας ζήτησαν να αυξήσουν το προσωπικό τους για να μπορούν καλύτερα να παρακολουθούν τη στατιστική κατάσταση στην Ελλάδα χωρίς με ένα ad hoc screening μπορέσαμε να φτάσουμε σε πολύ μικρότερη αύξηση του προσωπικού, 3% μόνο από ό,τι είχε αρχικά ζητηθεί. Χρησιμοποιούμε επίσης τα στοιχεία αυτά στην αναδιοργάνωση που χρειάζεται λόγω των νέων ε, χαρτοφυλακίων των επιτρόπων. DG Κλίμα, DG Ενέργεια, DG Κίνηση, DG Δικαιοσύνη, DG Εσωτερικά, Εσωτερικές Υπόθεσεις και προσέχουμε τις περιορισμένες διοικητικές δαπάνες για αυτές τις νέες γενικές διευθύνσεις. Και φυσικά εξετάζουμε πολύ προσεκτικά οποιοδήποτε αίτημα για αύξηση προσωπικού καθώς και το επίπεδο των διοικητικών δαπανών, που είναι πολύ σημαντικό. Για το μέλλον, έχουμε ένα πολύ σημαντικό έργο. Πώς θα να δημιουργήσουμε την Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τη νέα υπηρεσία, ε, διάφορες ε, συμφωνίες για τις αμοιβέ, ε, για την ασφάλεια, για την διοικητική στήριξη, για τη διοίκηση. Και πάλι θέλουμε να κάνουμε οικονομίες κλίμακας και να βοηθήσουμε την Κάθριν Άστον να ανταποκριθεί στη δέσμευσή της που λέει ότι θα πρέπει να αποδείξει ότι η νέα υπηρεσία θα επιφέρει 10% κέρδος και πιστεύω πως μαζί μπορούμε να το πετύχουμε. Ταυτόχρονα, και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω, οι προσπάθειές μας στον τομέα αυτό είναι περιορισμένες, γιατί όχι περιορισμένες, αλλά στην ουσία προσκλούν σε διάφορα εμπόδια, διότι διαρκώς ε, νέα αιτήματα, νέες προτεραιότητες μας έρχονται και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτά με την ανακατανομή του προσωπικού μας. Ε, ε, υπάρχουν δυνατότητες για περαιτέρω μείωση του κόστους σε συνεργασία με τις ε, ε, τους διάφορους οργανισμούς. Εγώ συνεργάζομαι με μια ομάδα για τις, τους οργανισμούς. Συμμετέχουν εκπρόσωποι από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και από την Κομισιόν φυσικά. Κάποια πιο, πιο επιφυλακτική στάση κρατούν τα κρατημέλη, αλλά σίγουρα είναι ένα τομέα όπου μπορούμε να κάνουμε πολλές οικονομίες. Και βέβαια, καλύτερο συντονισμός της δουλειά μας ε, χρειάζεται γιατί θα πρέπει να, να απασχοληθούν 50 ε, άτομα για να εξετάζουν τα έγγραφα τα οποία φτάνουν από το Κοινοβούλιο. Μέχρι στιγμής έχουμε λάβει 6.600 ερωτήσεις. Σημαίνει δηλαδή πολύ προσωπικό που ασχολείται με το να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις. Είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον όχι μόνο να αναζητήσουμε κέρδος αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους αλλά για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε το προσωπικό της ε, Κομισιόν να διατηρήσει την εμπειρογνωμοσύνη του, την ανταγωνιστικότητά του και την ισχυρή του διοικητική δυνατότητα, γιατί ε, το χρειαζόμαστε αυτό αν θέλουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που αναμένουν από εμά οι πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Επίτροπε. Αρχίζουμε τη συζήτηση. Αμέσως το λόγο έχει κυρία Γκρέσλα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Είναι μεγάλη ημέρα σήμερα. Σαν να έχουμε Πάσχα και Χριστούγεννα μαζί, γιατί σήμερα το Κοινοβούλιο για πρώτη φορά ασχολείται με τέτοια έλεγχο και η Κομισιόν κάνει τον έλεγχο αυτό του προσωπικού από το 2007 μετά από αίτηση του Κοινοβουλίου. Είναι λοιπόν έτοιμα της Επιτροπής μας. Μία φορά κάθε χρόνο ε, λαμβάνουμε την έκθεση αυτή και την τελευταία φορά ε, δεν είχα καν, ε, δεν κέρδισα καν ε, την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας δίνει τα στοιχεία αυτή. Και νομίζω ότι είναι υποδειγματικός ο τρόπος που δουλεύουμε. Η δίκησή μας εξετάζεται, περνάει από έλεγχο. Και γι' αυτό λοιπόν τα αποτελέσματα του staff screening πάντα είναι, προκαλούν έκπληξη. Θεωρώ ότι είναι ένα σύγχρονος τρόπος management και θεωρώ ότι σωστά κάνουμε και ασχολούμαστε σήμερα με το θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο για πρώτη φορά, ελπίζω όμως όχι για τελευταία, γιατί είναι, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα μέσα που έχει στη διάθεσή τους. Θα πρέπει λοιπόν να το ακολουθήσουμε αυτό ως πρακτική στο μέλλον. Να ξέρουμε πώς δουλεύει ο κόσμος στο ιστορικό μας. Πρώτη ερώτηση. Το contract agents, οι contract agents δεν θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο ε, staff screening. Δεύτερη ερώτηση. Τι θα γίνει, μάλλον ίδια ερώτηση, τι θα γίνει αν συμπεριληφθούν όλοι αυτοί οι contract agents. Ε, κατά δεύτερον, βλέπουμε πόσο καθυστερημένα και πόσο αργά εξαγάγουμε μαθήματα από το staff screening έχουμε 50% για διοικητικές δαπάνες. Το ίμιση. Το άλλο 50% ε, εργάζεται στον ε, επιχειρησιακό τομέα, το άλλο 50% ήταν 50% ήταν στα overheads, στις διοικητικές δαπάνες. Ε, οποιαδήποτε εταιρεία θα είχε φαλυρίσει. Προς τα πού οδεύουμε λοιπόν. Τρίτο ερώτημα. Αυτό που είπατε στο τέλος τι θέλουμε να αποδείξουμε, τι θέλουμε να καταδείξουμε με το staff screening. Είπατε σε ό,τι αφορά τις γενικές ε, διευθύνσεις. Ε, όταν βλέπουμε τι δεν μας αναφέρεται στο staff screening είναι τα εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή πόσα τμήματα ιδρύθηκαν, πόσες γενικές διευθύνσεις ιδρύθηκαν. Τι γίνεται λοιπόν από το 2004 και μετά, γιατί διαπιστώνω ότι όλο και πιο πολύ συρρυκνώνεται η διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε όλο και πιο πολλές ηγετικέ θέσεις, πιο πολλές από ό,τι ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 100 Μάλλον 48 ε, θέσεις Γενικού Διευθυντή έχει προβλέψει η Επιτροπή και τώρα έχουμε 100. Πότε θα επατρέψουμε στις 84 και πάλι είχατε θέσει αυτούς τους ε, στόχους, αυτούς τους αριθμούς ως όριο. Και τι κάνετε για να καταπολεμήσετε αυτή την, ε, τον κατακαιρματισμό της διοίκησης, γιατί νομίζω ότι δεν έχει νόημα να έχουμε όλο και πιο πολλούς αρχηγούς και όλο και λιγότερους Ινδιάνους. Αυτό που σπάει όλα τα ρεκόρ είναι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ε, πουθενά δεν μπορούμε να βρούμε μία υπηρεσία με τόσο λίγους υπαλλήλους, γιατί Γιατί τι γινότανε. Μα, μάλλον, ποιες είναι οι προτάσεις. Ένας διευθυντής προς έναν υπάλληλο. Είναι αναλογία αυτή. Πού θα καταλήξουμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για την παρουσίαση αυτή και για τη δυνατότητα που μας δώσατε να τα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ε, ε, Σόντεμπεργκ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ θερμά και τον Επίτροπο για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση του screening. Εγώ είχα δει από την ημερήσια διάταξη ότι υπήρχαν δύο στοιχεία σε αυτό το σημείο ο ένα ήταν ε, έλεγχο του προσωπικού και δεύτερο ήταν ο δεοντολογικό κώδικα για του επιτρόπου. Η κώδικα συμπεριφορά για του επιτρόπου. Ήταν ε, διπλό αυτό το σημείο. Εκτό αν μιλήσατε για τον κώδικα αυτό συμπεριφορά των επιτρόπων και ήμουν αφηρημένο εκείνη τη στιγμή. Ή ίσως δεν ήσταν τόσο αναλυτικός ως προς αυτό το δεύτερο τμήμα της ε, η σα διάταξη στο σημείο αυτό. Α, είπατε μετά θα αναφερθεί αυτό το θέμα. Οκ. Ο κύριος Γκέιρ. Τρει ερωτήσει για το Code of Conduct, για τον κώδικα διδαντολογία. Αλλά θα μα μιλήσετε πιο πολύ μετά. Να σα ευχαριστήσω καταρχά για τι παρουσιάσει αυτέ. Ω καινούριο στην Επιτροπή αυτή δεν έχω ασχοληθεί ακόμα με το θέμα αυτό, αλλά θεωρώ ότι Πρόκειται για ιδέες για την εσωτερική οργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί πολλές φορές αναφέρεται ότι σε ομάδες επισκεπτών ότι είναι αρκετά περιορισμένοι οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι αναλογούν σε λιγότερους από όσους απασχολούνται σε μια πόλη όπως η Κολονία, όπως το Μόναχο. Να σας ρωτήσω το εξής για τα overheads. Είπατε κύριε Αντιπρόεδρε ότι, ότι η Γενική Διεύθυνση συνυπολογίζεται στον υπολογισμό τα overheads. Οι εσωτερικοί δηλαδή συνεργάτες, οι εσωτερικοί υπάλληλοι. Αν όντως, όπως, όπως είπε η κυρία Γκρέσλε, η αναλογία είναι 50% η αναλογία, 50 προς 50, θα είχαμε προβλήματα. τότε όμως τα αριθμητικά στοιχεία μεμονωμένα, να σας ρωτήσω πώς ορίζετε τα overheads. γιατί ίσως αυτό να έχει αρνητικά αποτελέσματα, αρνητικές επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τους υπολογισμούς. Ίσως αυτό να μας διευκόλυνε ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επαφές μας και την παρουσίαση της κατάστασης προς τον κόσμο. Ευχαριστώ κύριε Στάς. Θα ήθελα να πω ότι θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο αυτό το εγχείρημα του Επιτρόπου να έχουμε μια επισκόπηση της κατάστασης και μας υπέδειξε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την αύξηση του προσωπικού του δεν είναι ιδιαίτερα οικονομικό και ότι υπάρχει αρκετό επιπλέον προσωπικό τα τελευταία χρόνια τα οποία απασχολείται. Άρα μας βάλατε λίγο στη θέση μας ε, και πετάξατε το μπαλάκι σε αυτό το παιχνίδι μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Σωστό είναι αυτό βέβαια, γιατί τέτοια θέματα δεν θα πρέπει να τη χάνουν υποκριτικής αντιμετώπισης. Είχα κάποιες ερωτήσει να κάνω για τον κώδικα ε, δεντολογία, αλλά από ό,τι κατάλαβα θα πάρετε το λόγο πιο μετά για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε την ε, πρωτοβουλία των πολιτών. Μιλάμε για 50.000 ε, υπογραφές πολιτών οι οποίες θα υποβληθούν προς εσάς. σχετικά με το πώς ε, οι πρώην επίτροποι μπορούν να ε, αποκτήσουν θέση στον ιδιωτικό κλάδο. Και ζητείτε από την Πρωτοβουλία των Πολιτών να ρυθμιστεί γρήγορα το θέμα αυτό, κατεπηγόντως μάλιστα. Μέσα Νοεμβρίου νομίζω θα λάβατε την αίτηση αυτή. Και θα ήθελα λοιπόν να σχολιάσετε και την πρωτοβουλία αυτών των πολιτών για τις 50.000 υπογραφές. Thank Σας ευχαριστώ. Καταρχήν, ευχαριστώ θερμά την κυρία Γκρέσλε, γιατί δική της ήταν η ιδέα και η πρωτοβουλία για τη συζήτηση αυτή στην Επιτροπή σας και το αμύωτο ενδιαφέρον τη και η συνεχής πίεση που μα ασκεί έχει αποφέρει καρπούς, γιατί είμαστε πολύ προσεκτικοί πια με τα στοιχεία που σα παρουσιάζουμε. Και είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στον τρόπο υπολογισμού των overheads αυτή της διοικητική ε, υποστήριξη και συντονισμού και των δαπανών. Και μάλιστα εκπονώντα αυτή τη μεθοδολογία δημιουργήσαμε και μια νέα τεχνογνωσία και φυσικά, όπω είπε η κυρία Γκρέσλε, η μεθοδολογία μα ενδιαφέρει και άλλα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Πολύ ευχαρίστω να τη μοιραστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, γιατί ίσω χρησιμοποιηθεί και από άλλου σε αντίστοιχε διαδικασίε screening. Σε ό,τι αφορά του συμβασιούχου, του contract agents, ίσω εκεί υπήρχε πρόβλημα με την ορολογία. Γιατί εγώ συμπεριέλαβα τους contract agents, τους συμβασιούχους ναι, γιατί έχουμε 6.000 ε, τέτοιου συμβασίουχους και όταν είπα 7.500 ε, προσωπικό αναφερόμουν σε όσους δεν έχουν σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά πολύ συχνά εργάζονται στα γραφεία της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια συμβάσεων που έχουμε με διάφορες εταιρείες είναι επιδοτήσει, πρόκειται για ερευνητέ ή για οι δήμονε ε, τεχνολογιών πληροφορική που παρέχουν υπηρεσίε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν κρύβουμε τίποτα με τα στοιχεία αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι υπάλληλοι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά προσφέρουν υπηρεσίε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την λειτουργία. Και ο αριθμό είναι μεγάλο, όπω σα είπα. Ε, είναι 7.500. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό ο αριθμό των συμβασίουχων. Όταν μίλησα για τα overheads, τη διοικητική υποστήριξη και το συντονισμό, είπα ότι καταφέραμε να μειώσουμε τον αριθμό των ε, υπαλλήλων από 19% ε, σε 15%. Οπότε όλο και περισσότερα καθήκοντα ανατίθεται σε συμβασιούχου, ιδιαίτερα όταν είναι επαναληπτικά αυτά τα καθήκοντα ή διοικητικά. Χρησιμοποιούμε του συμβασιούχου γιατί μα ε, στοιχίζουν πιο φθηνά. Σα το λέω ειλικρινά. Και έχουν και πιο ελαστικέ συμβάσει. Και αυτή είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίσαμε εξαιτία των δημοσιονομικών και άλλων περιορισμών. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τους συμβασίουχους στην κατηγορία αυτή όλο και περισσότερο. Τι θα συμβεί στο μέλλον. Σας υπόσχομαι ότι και εγώ προσωπικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί για να επανεξετάσει το θέμα των overheads, γιατί χρειαζόμαστε όλο και πιο αυτοματοποιημένη διαδικασία, όλο και πιο εκτεταμένη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και περισσότερα overheads στο μέλλον. Βέβαια, μας ενδιαφέρει και στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα όταν θα συζητηθούν τα νέα δημοσιονομικά μέσα και ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός και να δούμε πώς μπορούμε να πλουστεύσουμε το έργο μας και πώς να εκπονούμε τους δημοσιονομικούς ε, κανονισμούς ώστε και να προϋποθέτουν αυστηρό έλεγχο αλλά χωρίς ε, τόσο επαχθές γραφειοκρατικό ε, επαχθή γραφειοκρατικό φόρτο. Γιατί αυτό είναι που απαιτεί πολλά, πολλές δαπάνες και είναι μια μορφή που ακούμε πολύ τακτικά και από τα κράτη-μέλη αλλά και από τρίτες χώρες στις οποίες προσφέρουμε αναπτυξιακή βοήθεια. Θέλουμε να μειώσουμε λοιπόν αυτό το γραφειοκρατικό άκθος. Και σε ό,τι αφορά την, ε, τις ε, θέσεις management, έχουμε τώρα φτάσει στο 100, έχει δίκιο η κυρία Γκρέσλερ. Προσπαθούμε μετά την ε, ανάληψη των καθηκόντων από την Επιτροπή δημιουργήθηκαν νέε γενικέ διευθύνσει και τώρα βρισκόμαστε σε μια ενδιάμεση φάση. Προσπαθούμε να κατασταλάξουμε και γνωρίζω ότι ο αριθμός αυτός 100 είναι υψηλότερος από το στόχο μας, αλλά στο μέλλον και τις μελλοντικές προτάσεις για τις υψηλόβαθμες θέσεις το πρόβλημα θα μας απασχολήσει. Πάντως αυτό το αποτέλεσμα καταλήξαμε μετά από πολύ ε, δύσκολες συζητήσεις. Πάντως μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο και τώρα προσπαθούμε να προσαρμόσουμε και το μέγεθος και τα χαρτοφυλάκια κατά κάποιο τρόπο των Γενικών Διευθύνσεων στα χαρτοφυλάκια των Επιτρόπων. Θα ήθελα να απαντήσω τώρα και στον κύριο Ζόντεργαρτ και στον κύριο Στάις. Σε ό,τι αφορά τον κώδικα διοντολογίας των, επι των Επιτρόπων. Θα σα κάνω μια σύντομη παρουσίαση. Σα διαβεβαιώ πάντω ότι πήραμε πολύ σοβαρά τι υποδείξει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και τι παρατηρήσει των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί τώρα έχουμε και την πρωτοβουλία των πολιτών και θα εξετάσουμε πολύ σοβαρά όλε τι συστάσει. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια του κ. Γκάιερ για την αξιολόγηση των καθηκόντων και τα θέματα επικοινωνίας. Δίκιο έχετε κύριε Γκάιερ ότι μερικές φορές παραείμαστε αυστηροί και απαιτητικοί με τους εαυτούς μας. Αλλά μας ενδιαφέρει να είμαστε σχολαστικοί, αυστηροί, ακριβείς και ταυτόχρονα να δούμε ποια είναι τα καθήκοντα των Γενικών Διευθύνσεων και συγκεκριμένων μονάδων σε μια εξελικτική διαδικασία. Γιατί όσο αναλαμβάνουμε περισσότερα πολιτικά καθήκοντα, είναι σαφές ότι θα πρέπει ε, μερικοί από τα overheads να πάνε σε άλλες δραστηριότητες, από διοικητικά καθήκοντα σε πιο πολιτικά, οπότε θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ακριβής ορισμός αυτού του overhead, διοικητική υποστήριξη και συντονισμός και ποια είναι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των frontline activities και των διοικητικών ε, δραστηριοτήτων. Πάντως ε, σας υπόσχομαι ότι δεν πρόκειται να κάνουμε κανένα κόλπο ή κανένα τέχνασμα, θα σας ενημερώνουμε τακτικά Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε υπό στενό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα σας ενημερώσουμε για τις μετακινήσεις από τη μία μονάδα στην άλλη. Και θα καταφέρουμε, πιστεύω, να σας πείσουμε για τη λογική όλων αυτών των μεταθέσεων. Και για τα θέματα επικοινωνίας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε στο μέλλον τα overheads ε, όσο γίνεται πιο πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ε, εισήγησή σας και δίνω το λόγο στην κυρία Γκρέσλα. Να σας υπενθυμίσω απλά ότι σε ό,τι αφορά το screening πρόκειται για ε, απόρρια της ε, μεταρρύθμισης της διοίκησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί υπάρχουν γενικές διευθύνσεις όπως η προϋπολογισμού, διοικητική, ε, γλωσσική κτλ. Και κάθε γενική διεύθυνση έχει ε, υποτμήματα. Άρα η διέρεση σε υποτμήματα, αυτό αποτέλεσε την αιτία του εγχειρήματο αυτού. Για να δούμε πού μπορούμε να απλοποιήσουμε τις εργασίες μας. Αυτό τι σημαίνει. Ότι θέλουμε να δούμε τι συμβαίνει στις κάθε γενικές, στην κάθε γενική διεύθυνση και τα συμπεράσματα τα οποία εξαγάγονται θα πρέπει να λάβουν συνέχεια. Γιατί βλέπω ότι οι κεντρικές γενικές διευθύνσεις αυξάνεται ε, η στελέχωση, αντιναμιώνεται. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε γιατί συμβαίνει αυτό. Πρόκειται για έναν αιώνιο αγώνα ε, στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταξύ κεντρικής και απόκεντρης ε, ε, διαμόρφωσης, διαρρύθμισης των εργασιών. Είναι σημαντικό για μας να δούμε πώς εφαρμόζεται, για παράδειγμα, ε, η νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Θέλουμε να υπάρχει πιο έντονο έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη. Δεν έχω την εντύπωση ότι το θέμα αυτό ε, την χάνει τη αντίστοιχη προσοχή που θα έπρεπε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, είναι πολύ περιορισμένο για παράδειγμα ο αριθμό ατόμων που ε, ελέγχουν την εφαρμογή των περιβαλλοντικών προτύπων στα κράτη-μέλη. Μπορείτε να μα πείτε λοιπόν πόσοι ακριβώς ε, ασχολούνται με την παρακολούθηση της κοινωτικής νομοθεσίας και της εφαρμογής αυτής στα κρατημέλη. Θα μας βοηθούσε αυτό. Παρακαλώ, μπορούμε... μπορείτε να απαντήσετε και μετά να περάσετε στο δεύτερο τμήμα. Να απαντήσω στην κυρία Γκρέσλε. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Γκρέσλε, ότι όταν ελήφθη η απόφαση για την αποκέντρωση ήταν πολύ σωστή για τη γενικέ διευθύνσει ήταν σαφέ ότι θα χρειαζόταν ένα περιθώριο κινήσεων και λιγμών, μια αυτονομία για να είναι και πιο αποτελεσματικέ. Και η διαδικασία αποκέντρωση ήταν πολύ σημαντική και πολύ εύστοχη από άποψη διαχείριση. Βέβαια, νομίζω ότι το παρατραβήξαμε τελικά με την αποκέντρωση, γιατί ως ιδέα ήταν σωστή, αλλά ίσως ήταν υπερβολικό αυτό που έγινε. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη τεχνολογία πληροφορικής, αυτό το κλάδο στην Επιτροπή. Εκεί οι γενικές διευθύνσεις αποφάσισαν να αναπτύξουν τα δικά τους συστήματα που θα ήταν κομμένα και ραμμένα για τα δικά τους μέτρα. Οπότε καταλήξαμε σε μια κατάσταση να έχουμε πολλά συστήματα, πληθώρα συστημάτων που δεν είναι εύκολο να επικοινωνούν μεταξύ τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση στο θέμα της πληροφορικής θα χρειαζόμαστε και ένα συντονιστικό σώμα, ένα φορέα που θα συντονίζει τι γίνεται, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα πληροφορικής, ώστε οι providers να ξέρουν τι περιμένουμε από αυτούς, να μην υπάρχουν επικαλύψεις και να έχουμε και μία ε, ε, καλύτερη εμπειρογνωμοσύνη και τη δυνατότητα να, αφισβητούμε να και τα αιτήματα μερικών γενικών διευθύνσεων για συγκεκριμένα προγράμματα. Αυτά συνέβησαν ως προς το τομέα της πληροφορικής. Ήδη έχουμε μια νέα δομή διακυβέρνησης για τις τεχνολογίες πληροφορικής με την, το ABM συν IT Group διασφαλίζοντας ένα καλύτερο συντονισμό, ένα συντονισμό σε υψηλό επίπεδο προκειμένου να υιοθετούμε πιο συλλογικές λύσεις και για το θέμα του, της πληροφορικής αλλά και το θέμα των ε, ε, ανθρωπίνων πόρων, του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί χρειάζεται αυτό όχι μόνο στην πληροφορική, αυτός ο συντονισμός, αλλά και στους ανθρώπινους πόρους. Το, το κοινωτικό δίκαιο είναι ε, εκτενές αυτά τα θέματα και υπάρχουν βέβαια διαφορές στα κράτη-μέλη και διαφορετικός βαθμός εφαρμογής. Πάντως, αν δείτε το ποσοστό του προσωπικού ή τον αριθμό των υπαλλήλων που ασχολούνται, για παράδειγμα, με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, θα το ψάξω και θα σας δώσω τις σχετικές πληροφορίες. Ευχαριστώ. Και τώρα να περάσουμε στο δεύτερο σημείο της της διάταξης, που είναι ο κώδικας διοντολογίας των επιτρόπων. Ξέρω ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ενδιαφέρει την Επιτροπή σας. Και επίσης γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να βάλει σε αποθυματικό τα έξοδα τα δικητικά για το 2011. Μέχρι ότου υπάρχει πολιτική δέσμευση εκ μέρους μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αναμένεται να υποβάλει έναν μεταρρυθμισμένο κώδικα δεντολογίας μέχρι τα τέλη του έτους. Θα ήθελα λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό θα συμβεί σε κάθε περίπτωση και να σας ενημερώσω ότι ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε στην την αναθεώρηση του κώδικα δεντεολογίας αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας πλαισίου. Γιατί περιμέναμε μέχρι τη στιγμή αυτή όμως, γιατί ξέρετε ότι οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία πλαίσιο ήταν αρκετά περίπλοκες και όλα τα θεσμικά όργανα ήταν πολύ ενθουσιασμένα με τον τρόπο που διεξήχθησαν οι διαπραγματεύσει. Θέλαμε λοιπόν να ολοκληρωθεί καταρχά η συμφωνία όχι Χάρηκα που ήταν τόσο καλή η συμφωνία αυτή που υπεγράφει. Από αυτή τη στιγμή λοιπόν και μετά ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε και να κοιτάμε τον κώδικα δεοντολογίας. Δεν είμαι απόλυτα ακριβής, θα θα με επιτρέψετε, θα με συγχωρήσετε, γιατί ο πρόεδρός μας ζήτησε από όλους τους επιτρόπους να υποβάλουν προτάσεις για την βελτίωση του κώδικα. Και η προθεσμία καταλεκτική ήταν η προηγούμενη Παρασκευή για την υποβολή των προτάσεων αυτών. Άρα, ο κώδικας διοντολογίας θα συζητηθεί στις 18 Νοεμβρίου προβλέπεται και αναμένω ότι πολύ σύντομα μετά από τις συζητήσεις αυτές μεταξύ των επιτρόπων θα υποβληθούν τα συμπεράσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να είμαι πιο συγκεκριμένο, ποιε θα είναι οι κατευθυντήριε γραμμέ. Θα θέλουμε να βελτιωθεί ο κώδικα διαιτολογία, να διευκρινιστούν τα θέματα τα οποία τίθενται συχνά από το κοινό και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και φυσικά, επειδή είμαστε ε, υποχρεωμένοι να σεβόμαστε τις ε, συνθήκες. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι ανεξάρτητα, δεν θα πλήττονται από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων και ότι θα υπάρχει αξιοπρέπεια και ευχέρεια. Τα θέματα λοιπόν αυτά όλα θα τα εξετάσουμε και θα εξετάσουμε το πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε στα πιο συχνά ερωτήματα. Αυτά λοιπόν τα θέματα σχετίζονται με το πώς ε, οργανώνονται οι πολιτικές δραστηριότητες των επιτρόπων, πώς μπορούμε να ε, αναδιοργανώσουμε τη σύγκρουση συμφερόντων και την ε, διανομή των συμφερόντων των επιτρόπων, πώς θα πρέπει να ρυθμίζουμε τις δραστηριότητες των επιτρόπων μετά το τέλος της θητείας τους και πώς μπορούμε να διευκρινίζουμε τους κανόνες για τη φιλοξενία. Αυτά είναι λοιπόν τα θέματα τα οποία μας απασχολούν και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με τις ε, υπηρεσίες για να βρούμε τις λύσεις που θεωρώ ότι θα γίνουν αποδεκτές κατά μεγάλο βαθμό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις οποίες ελπίζω ότι θα ε, εγκρίνει το Κολέγιο των Επιτρόπων μέχρι τις 18 του μηνός. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές δραστηριότητες, η Επίτροπη που θέλουν να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές θα πρέπει να τηρούν κάποιες βιογραφές πριν το τέλος της προηγούμενης ε, εθνίας. Και θα ορίζεται ποιο μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αναλάβει τις αρμοδιότητές τους από το σημείο αυτό και μετά. Και το ίδιο ισχύει και σε πολιτικές δραστηριότητε για τις εθνικές εκλογές. Τώρα, Γνωρίζω ότι υπάρχουν αιτήματα για την παράταση της περίοδου κατά την οποία οι πρώην επίτροποι θα πρέπει να ειδοποιήσουν την Επιτροπή για τις, τέτοι... για τις τους αυτές. Θα θέλαμε να καταστεί απόλυτα σαφές ότι οι επίτροποι δεν πρόκειται να κάνουν λόμπι, ούτε θα υποστηρίξουν, ε, ούτε θα κάνουν συναντήσεις με μέλη της Επιτροπής ή με προσωπικό της Επιτροπής, με πελάτες και ούτω καθεξής, ε, οι οποίοι κινούνται στο πλαίσιο των πρώην αρμοδιοτήτων τους. Νομίζω ότι είναι σαφές λοιπόν τι είδους συμπεριφορά μπορούν να επιδείξουν οι επίτροποι σε ό,τι αφορά με τους, τους πρώην υπαλλήλου, τους πρώην συναδέλφους τους. Ένα άλλο θέμα, η δήλωση συμφερόντων. Συμφωνώ στο σημείο αυτό μαζί σας ότι ασκήθηκε έντονη κριτική ότι η δήλωση των συμφερόντων δεν ενημερώνεται αρκετά συχνά και θα τις συμπεριλάβουμε στον κώδικα διολογίας. Θα πρέπει τακτικά να ενημερώνεται η δήλωση συμφερόντων. Να είναι πιο διαφανής, πιο ευανάγνωστη. Θα πρέπει να περιέχονται όλα τα στοιχεία τα οποία μπορούν να στοιχειοθετήσουν σύγκρουση συμφερόντων, για παράδειγμα κατοχή μετοχών εταιρεία. Και επίσης θα συμπεριληφθούν και οι σύζυγοι αλλά και οι σύντροφοι των επιτρόπων. Αυτό φυσικά ελπίζω ότι θα συνεισφέρει στην περαιτέρω διαφάνεια και στην περαιτέρω σαφήνεια των δραστηριοτήτων των επιτρόπων. Επίσης, ένα άλλο συχνό ερώτημα. Τι συμβαίνει αν ένας επιτρόπος ε, αντιμετωπίσει σύγκρουση συμφερόντων. Είναι σαφές ότι αν τέτοιο περιστατικό παρουσιαστεί, το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκι, το συγκεκριμένο θέμα θα εκχωρηθεί σε άλλον επίτροπο και θα ειδοποιηθεί άμεσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προσωπία στο εξωτερικό και πάλι στα σταφές ότι οι επίτροποι ε, ακολουθούν τους ίδιους κανόνες όπως και το υπόλοιπο προσωπικό της Επιτροπής, δηλαδή ότι σεβόμαστε πλήρως τους χρηματοοικονομικούς κανονισμούς και τους κανόνες εφαρμογής του γενικότερου προϋπολογισμού της Ένωσης και πάλι λοιπόν δεν υπάρχει οποιαδήποτε αφησιμία. Τώρα, επικρίσεις για το προσωπικό των επιτρόπων, των γραφείων των επιτρόπων. Εξετάσαμε τι γίνεται και αλλού και θα συμπεριληφθούν νέες διατάξεις ότι γενικά οι σύζυγοι, οι σύντροφοι και τα άμεσα μέλα της οικογένειας των επιτρόπων δεν μπορούν να απασχολούνται στα γραφεία τους. τρία τελευταία σημεία σε ό,τι αφορά τις δωρεές. Γιατί ξέρετε ότι στον κόσμο της διπλωματίας ε, δεν είναι ασυνήθιστο να γίνονται δώρα. Θα διευκρινιστεί ότι ο Επίτροπος δεν μπορεί να δέχεται δωρεές πάνω των 150 ευρώ. Δώρα πάνω από 150 ευρώ σε ό,τι αφορά θέματα φιλοξενία, Προσπαθούμε να διευκρινίσουμε τον κανόνα, τους κανονισμούς με τέτοιο τρόπο, ώστε σε περίπτωση φιλοξενία, η οποία προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων δεν θα μπορεί να γίνεται δεκτή η φιλοξενία αυτή προκειμένου να μην δίνεται η εντύπωση καν ότι μπορεί να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Επιτρέψτε μου να μιλήσω για την ε, Δεντολογική Επιτροπή. Θα ξέρετε ότι ως τώρα η Επιτροπή Διεντολογίες ε, εργάζονται ως Επιτροπή Ad Hoc. Θα θέλαμε να βελτιώσουμε όμως τις εργασίες της Επιτροπής αυτής για το μέλλον. Άρα εξετάζουμε το ενδεχόμενο να διευρύνουμε την Επιτροπή Διεντολογίας και εξετάζουμε το ενδεχόμενο εισαγωγής ε, επιπρόσθετων στοιχείων. Καταρχάς, όταν η Επιτροπή Διεντολογίας καταλήξει στο συμπέρασμα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο χύψη επίτροπος μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντά του. Είμαι βέβαιος ότι αυτό... μάλλον θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωρίζει πώς κατέληξε στο συμπέρασμα αυτά, αυτό η Επιτροπή Δεντεολογίας, με ποια συμπεράσματα, με ποια επιχειρήματα. Και το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που καταλήξει σε αρνητικό συμπέρασμα η επιτροπή αυτή. Σε περίπτωση που καταλήξει το συμπέρασμα ότι ο Επίτροπο δεν μπορεί να λάβει τα καθήκοντά του. Θέλουμε να δημοσιεύονται τα αποτελέσματα αυτά για να υπάρχει διαφάνεια τη Επιτροπή αυτή. Επιπλέον, θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή Διεντολογία να ε, προετοιμάζει τακτικές εκθέσεις, μία κάθε πενταετία τουλάχιστον, που θα παρουσιάσονται ε, στο μέσο της θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι στο τέλος, στο μέσο της θητείας της, μία έκθεση για το πώς ε, οι αρχές διεντολογίας ε, γίνονται σεβαστές και πώς τηρούνται οι σχετικές διτάξεις. Συνοψίζοντας, κύριε Πρόεδρε, ελπίζω η Επιτροπή σας να με συγχωρέσει που δεν, μπορεί, δεν μπορώ να επισέλθω σε περισσότερο λεπτομέρειες. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η σημερινή κατάσταση και θα αποφασίσουμε πιο πολλά στις 18 Νοεμβρίου. Όταν θα γίνει αυτό, φυσικά θα ενημερωθεί άμεσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τελευταία πρόταση που έχω να πω Εργαζόμαστε σκληρά για τον κώδικα δεντολογίας των επιτρόπων, αλλά έχουμε πει και στο παρελθόν ότι δεν ήταν κακή ιδέα να υπάρχει αυτός ο κώδικας δεντολογίας ως, ε, μια, ως ένα σημείο αναφοράς για ένα διαθεσμικό κώδικα δεντολογίας για το πώς αντιμετωπίζουμε θέματα διαφάνειας. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια καλή ιδέα και την οποία θα πρέπει να συζητήσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Χατζη Μαρκάκης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την πολύ επιτυχία αυτή παρουσίαση. Χαίρομαι που δίνεται τόσο ιδιαίτερη σημασία στην Επιτροπή Διδεολογία. και πραγματικά θεωρώ ότι είναι καλό να υποβάλει τακτικά εκθέσεις. Να θίξω ένα σημείο το οποίο ως τώρα ήταν λίγο διαφορετικό. Το θέμα της δήλωσης συμφερόντων. Κοιτώντας την έκθεση των ε, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις στον τομέα αυτών. Γι' αυτό λοιπόν πολλοί ευρωβουλευτές έχουν την εντύπωση ότι ε, εξηγούν και δημοσιεύουν την οικονομική τους κατάσταση, το οποίο είναι σωστό, αλλά αναμένουμε το ίδιο να συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε μια ετήσια αναθεώρηση. Εμείς μάλλον κάθε χρόνο ε, δηλώνουμε τα οικονομικά μας συμφέροντα, το οποίο ποτέ δεν γίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ω τώρα. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι που προβλέπετε και μια τακτική τέτοια υποβολή των συμφερόντων. Αλλά δεν είναι Για παράδειγμα το γεγονός ότι υπάρχουν πέντε επιτροποί οι οποίοι δεν ικανοποιούν αυτές τις ε, διατάξεις. Υπάρχει επίσης και το θέμα των κενών θέσεων και των ε, θέσεων ε, χωρίς αμοιβή. Όλα αυτά θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Μία ερώτηση έχω να σας απευθύνω. Μιλάμε για τη σκέψη να δημιουργηθεί ένας κώδικας δεντολογίας το, οποίο οποίος θα αποτελούσε βάση για όλα τα θεσμικά όργανα. Με τον κύριο Φανρόμπαϊ έχουμε και μια, ένα νέο θεσμικό όργανο από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ένα νέο θεσμικό όργανο τον οποίο, του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα δεν τα έχω δει πουθενά. Το ίδιο ισχύει και για την Αντιπρόεδρο, την Λέδη. Άστον υπάρχουν πλέον νέα θεσμικά όργανα όπου θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας κοινό κώδικας διοντολογίας. Εμείς ως Κοινοβουλίο έχουμε προχωρήσει αρκετά. Ναι, οκ, okay, μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα ε, ως ένα βαθμό. Αλλά ποια είναι η θέση σας σε ό,τι αφορά έναν κοινό κώδικα διοντολογίας. Θα ήθελα να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ κύριο Σόντεργαρτ. Όχι, έναν Ευχαριστώ για τα θέματα διαφάνειας. Φυσικά, όπως είπατε και εσείς, ένα θέμα είναι η διαφάνεια σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Δεντολογίας, αλλά από την άλλη υπάρχει και θέματα α, σε ό,τι αφορά την ε, νέα απασχόληση πρώην επιτρόπων, για την οποία θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή. Το ερώτημά μου που αφορά τη διαφάνεια είναι το εξής. Μήπως θα μπορούσαμε να, θέσουμε πιο, να δώσουμε πιο πολύ διαφάνεια σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τη δημοσίευση τέτοιων πληροφοριών στο διαδίκτυο. Ναι, αν θα μπορούσατε, λέει ο Επίτροπος, να επαναλάβετε το πρώτο τμήμα της ερώτησής σας σε ό,τι αφορά την δημοσίευση των νέων θέσεων πρώην επιτρόπων. Πρέπει να, να αναφέρουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις νέες τους δραστηριότητες. Και εδώ χρειάζεται πιο πολύ διαφάνεια, γιατί προηγουμένως είπατε ότι χρειάζεται μόνο μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις εργασίες της Επιτροπής Διαντολογίας αλλά σε ό,τι αφορά την διαδικασία Έγκριση αν θέλετε, των νέων θέσεων των επιτρόπων, θεωρώ ότι και εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Ποια είναι η δική σας θέση, λοιπόν, ρωτώ. Η συνάδελφος Γκρέσλα. Ευχαριστώ. Να πω το εξή. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη με αυτά που προφορικά μας αναφέρετε αυτή τη στιγμή, αλλά να περιμένω να δω τι θα μας πείτε και γραπτά. Τι θα μας υποβάλλετε γραπτά. Γιατί Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι εμπιστευτικά και απόρριτα όλα αυτά τα θέματα. Δημόσια θα πρέπει να είναι. Και χαίρομαι που συγκεντρώσαν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις 200.000 υπογραφές για την διαφάνεια αυτή. Δεν θα πρέπει να απογοητεύσουμε την κοινή γνώμη. Κοιτώντας ε, τις ε, δημοσιονομικές ε, δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τι να πω, κακομίτιδες. Κάτι δεν πάει καλά. Γιατί αν έχετε τόσα λίγα, πολύ λυπάμαι, γιατί όλοι οι πολιτικοί είμαστε και έχουμε εργαστεί, έχετε εργαστεί μια ολόκληρη ζωή. Ε, μα είναι δυνατόν να έχω εγώ πιο πολλά από εσά, τι να σας δανείσω. Έχω λοιπόν πάρα πολύ μεγάλες αμφιβολίες και κοιτώντας λοιπόν και τις ε, χρηματοοικονομικές δηλώσεις έχετε κάνει και ένα λάθος για τους νέους κανόνες. Δεν θεωρώ ότι θα ήταν καλή ιδέα να μην ρυθμιστούν τα μεταβατικά κονδύλια. Αυτό φυσικά δεν είναι πολύ απλό και το ξέρουμε, το έχουμε συζητήσει. Υπάρχει και σχετική απόφαση του Συμβουλίου. Γιατί ένα υπουργό εξωτερικών Ιταλία θα πρέπει να λαμβάνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή είχε υπάρξει ε, στο παρελθόν επίτροπος. Γιατί θα πρέπει και τα, τα ευρωπαϊκά, τα, τα μέλη του ε, Κοινοβουλίου να παίρνουν λεφτά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι πάει να πει αυτό, όποιος έχει αφήσει μια θέση την έχει αφήσει. Δεν μου αρέσει αυτό σαν ιδέα να υπάρχουν τέτοια μεταβατικές ε, αμοιβέ. Θα πρέπει λοιπόν να το διευκρινίσουμε αυτό και ξέρω ότι όλα αυτά δεν πρέπει να σας κάνουν πιο αγαπητό μεταξύ των συναδέλφων σας. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώς μπορούμε, θα ήθελα μάλλον να τονίσω ότι θέλουμε ένα καθαρό κώδικα δεντεολογίας και να λάβουμε υπόψη και το κίνδυνο να μας βγει η φήμη. Όλο τον έχουμε τον κίνδυνο αυτό, ιδιαίτερα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί είναι μεγάλη παγίδα. Είναι ίσως η μεγαλύτερη παγίδα που έχουμε μπροστά μας οι βουλευτές έχουν λάβει μια εντολή από τον κόσμο και αυτό είναι μια βασική διαφορά από τους επιτρόπους. Δεν είναι δυνατόν, ούτε είναι καλή ιδέα να προσπαθήσουν οι επίτροποι λοιπόν να αφήσουν αυτό το θέμα και να το βάλουν κάτω από το χαλί. Η ιδέα του να υπάρχει ένας κανόνας για όλους. Όμως θεωρώ ότι δεν είναι σωστή ούτε δέουσα. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Να μιλήσω για αυτή τη διαφορά που έκανε η κυρία Γκρέσλε, ότι είμαστε δηλαδή ε, άτομα, ότι έχουμε εντολή του από το λαό. Όντως έτσι είναι. Χάρηκα με αυτά που μας είπε ο Επίτροπος. Αλλά όντω αυτά είναι προφορικά. Και πολύ συχνά πρέπει να δούμε τέλο πάντων τι θα γίνει και με τα έγγραφα που θα λάβουμε. Σε τέτοια αφορά τα θέματα αυτά, σίγουρα δεν θα είστε πλέον αγαπητός ε, μεταξύ των συναδέλφων σας. Θεωρώ λοιπόν ότι θα λάβετε την υποστήριξη όλη τη κοκομπού και τι να κάνουμε και εμεί ω Επιτροπή δεν είμαστε πλέον αγαπητοί του Κοινοβουλίου. Αλλά θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπε στο τέλο η κυρία Γκρέσλε. Θα ήθελα να υποδείξω το εξή. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τον Επίτροπο σε ό,τι αφορά την βελτίωση τη τρέχουσα νομοθεσία, σε ό,τι αφορά τον κώδικα θεντολογία των επιτρόπων, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε ότι και εδώ στο Κοινοβούλιο υπάρχουν πολλά τα οποία δεν είναι τέλεια. Σας άκουσα κυρία Γκρέσλε στα γερμανικά. Μιλήσατε για κακομύριδες. Κοιτώντας ε, τις ε, οικονομικές δηλώσεις των επιτρόπων ότι υπάρχουν πολλοί κακομύριδες. Πολλοί και στο Κοινοβούλιο είναι κακομύριδες. Κοιτώντας ε, την ιστοσύλληλα το, του Κοινοβουλίου και τις ε, οικονομικές δηλώσεις των συναδέλφων και τι λένε ότι κερδίζουν, τι, τι λένε ότι βγάζουν και κοιτώντας τι γίνεται και στην πράξη, ε, νομίζω ότι και εδώ υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ και στον κύριο Ιτάλα που είναι ε, εισηγητής ε, για την απαλλαγή. Υπάρχει όντως η διαφορά αυτή που λέτε μεταξύ βουλευτών, αρετών βουλευτών και των επιτρόπων. Αλλά νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό αυτή η άσκηση να γίνει και για το συντορικό του Κοινοβουλίου, για να δούμε ποια είναι η αντιμετώπιση του κόσμου ως προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτό. Αυτό που κάνετε, αυτό που γίνεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να γίνει και για το Κοινοβούλιο. Χωρίς να μπουν όλα στο ίδιο καλάθι και να χαθούν οι διαφορές. Θα πρέπει να συμβούν και τα δύο. Και οι δύο αυτές ασκήσεις. Ο Στάλφος Αγαπητέ κύριε Στάς, συμφωνώ όταν λέτε ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και τα δικά μας και τα, τα του μου οίκου. Χαίρομαι με αυτά που άκουσα για τη βελτίωση του κώδικα τεντεολογίας. Μία διάμεση παρατήρηση. Ένας ε, υπάλληλος μας είχε μιλήσει στην αρχή της θητείας μου για τον Μπαρόσο. Καταλαβαίνουμε φυσικά, Επίτροπε, ότι υποβάλλοντας τέτοιες προτάσεις δεν θα είστε αγαπητός μεταξύ των συναδέλφων σας, αλλά θέλουμε σαφήνεια, θέλουμε διαφάνεια. Αν ε, τηρήσετε τις αρχές αυτές, θα έχετε ως σύμμαχο την Επιτροπή μας και στο σημείο αυτό. Θέλουμε μια Ευρώπη η οποία θα έχει καλή φήμη ανεξάρτητα αν πρόκειται για επιτροπή, για βουλευτές, για υπαλλήλους. Ας τα βάλουμε αυτά σε ένα καλάθι. Να μην έχει τη φήμη η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι κοιτάει μόνο τα δικά της συμφέροντα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε λοιπόν σαφείς κανόνες, διαφάνεια. Και να λέμε ότι κοιτάξτε αν θέλετε τα στοιχεία αυτά και να εξετάσετε εσείς οι ίδιοι αν ισχύουν αυτές οι κατηγορίες που ακούτε. Αυτό μόνο με διαφάνεια μπορούμε να το πετύχουμε. Να πω δύο λόγια τώρα για αυτές τις αμοιβέ τις μεταβατικές. Ένας υπάλληλο. θα πρέπει να έχει κάποιο χρόνο στη διάθεσή του μέχρι ότου βρει μια νέα θέση. Αυτό είναι ο σκοπός, φαντάζομαι. Ο μισθός ενός Επιτρόπου, ο οποίος λαμβάνει μια νέα θέση, προστίθεται στον προηγούμενο μισθό του. Τι κίνδυνος ε, ελοχεύει. Ε, σε περίπτωση που υπάρχει κάποια μέγιστη περίοδος ε, τέτοιου μεταβατικού μισθού να κατηγορηθεί ο, επίτροπος, ο πρώην Επίτροπος ότι πρόκειται για άεργο. Δεν γίνονται λοιπόν αυτά σε ό,τι αφορά την συσσόρευση και ε, το άθροισμα των μισθών ενός επιτρόπου, για παράδειγμα. Αυτές είναι οι δικές μου κόκκινες γραμμές. Να κάνω και εγώ μια τελευταία παρατήρηση και μετά δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο. Η Κομισιόν σκέφτεται να συντάξει ένα νέο κείμενο με παραπομπή σε οποιαδήποτε περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων όπως μπορεί ας πούμε να προκύψει ε, μεταξύ της θέσης ενός επιτρόπου και οποιαδήποτε άλλης, ε, από οποιοδήποτε άλλο λειτουργήματος. Πώς μπορούμε δηλαδή να εγγυηθούμε την ανεξαρτησία του επιτρόπου σε σχέση με τη χώρα προέλευσης που τον διόρισε. Θα, θα θυμάται ο Επίτροπος ε, Σιεύκοβιτς ότι εγώ έκανα μία μια τέτοια ερώτηση κατά τη διάρκεια της ακρόασης σε σχέση με τέτοια σύγκρουση συμφερόντων για κάποιον επίτροπο. Και έπειτα, πώς μπορεί να προχωρήσει στον διορισμό των μελών του επιτελείου του και εάν αυτή υπόκειται στους όρους που υπόκειται και οι υπόλοιποι πάλι της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις με τη σειρά που τέθηκαν. Κύριε Χατζημαρκάκη, έχετε απόλυτο δίκιο ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε το έργο της Επιτροπής Διαντολογίας και φυσικά να βελτιώσουμε τη διαφάνεια των σχέσεων και με τους πρώην επιτρόπους να υπάρχει διαφάνεια ως προς το κοινό και ως προς τις, υπόλοιπου, στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Για να είναι εξασφαλισμένη διαφάνεια της απόφασης κάθε επιτροπής ιδεοντολογίας. Για να ξέρει και ο πολίτης πού στηρίζεται η συγκεκριμένη απόφαση, άσχετα με το αν είναι θετική ή αρνητική. Να γνωρίζει πώς έγινε η ανάλυση, να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στις εργασίες της Επιτροπής Διοντολογία. Αυτή άλλωστε θα είναι μία από τις προτάσεις που θα κατατεθεί. Συμφωνώ με τους ε, ευρωβουλευτές ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα της δήλωσης συμφερόντων, γιατί όλοι καταθέσαμε δήλωση συμφερόντων λίγο πριν αναλάβουμε τα καθήκοντά μας ως Επίτροποι. Και οι δηλώσεις αυτές είναι πλήρεις, αλλά Τώρα θέλουμε να αποσαφηνίσουμε αυτό το θέμα, να συμπεριλάβουμε και τους συντρόφους και συζύγους, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι τώρα, δεν καλύπτονταν οι σύζυγοι και οι σύντροφοι από τις δηλώσεις συμφερόντων και επίσης να είναι σαφές που μπορεί να βρει κανείς αυτές τις πληροφορίες, γιατί υπάρχουν μεν, αλλά πολύ συχνά είναι δυσπρόσιτε. Οπότε καλό θα ήταν να υπάρχει ε, ένας ε, ομοιόμορφος σύνδεσμος, ένα link όπου μπορεί κανείς να βρει τις δηλώσεις συμφερόντων συγκεκριμένων των επιτρόπων του που τον ενδιαφέρει. Ε, επίσης, ε, είναι απαραίτητη και μια τακτική ενημέρωση αυτών των δηλώσεων συμφερόντων. Δεν μπορεί να γίνεται άπαξη δήλωση και να μην υπάρχει συνέχεια. Και ε, καλό θα ήταν αυτέ οι ενημερωμένες δηλώσεις συμφερόντων να περιλάβονται στις δηλώσεις της χρηματοοικονομικές που παβάλλουν οι Επίτροποι. Όπως είπε η κυρία Γκρέσλερ, δεν είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει μια ενιαία ομοιόμορφη λύση για όλα τα θεσμικά όργανα, αλλά για την περίπτωση του κώδικα δοντολογία, καλό θα ήταν να εξετάσουμε και μια ομοιόμορφη εφαρμογή του. Ή κάτι παρόμοιο τουλάχιστον ε, προσπαθώ να κάνουμε με το Μητρό Διαφάνεια. Εκεί υπάρχει πολύ αγαστή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Και μέχρι στιγμή είχαμε πολύ θετικέ αντιδράσει και από το Κοινοβούλιο αλλά και από το Συμβούλιο, ότι είναι και το Συμβούλιο έτοιμο να ε, εξετάσει από κοινού μαζί μας το θέμα της διαφάνειας ε, των ε, διαφόρων λόμπι συμφερόντων. Γιατί νομίζω ότι είναι συμβολική αυτή η συνεργασία μεταξύ των κοινοτικών θεσμικών οργάνων για θέματα διαφάνειας. Επίσης, Είμαι βέβαιος ότι αν δοθεί μια διοργανική διάσταση σε αυτά τα θέματα θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα και από το ευρύ κοινό. Περιμένουμε λοιπόν μια κοινή συζήτηση για τα θέματα αυτά. Κύριε Ερενχάουζε, τι συμβαίνει με τους πρώην επιτρόπους και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και ποιο είναι το έργο της Επιτροπής Θεατολογίας για τα θέματα αυτά. Και εγώ το είχα αναφέρει βέβαια σήμερα αν ένας πρώην επίτροπος ενδιαφέρεται για μια νέα θέση, του προσφέρεται μια νέα θέση, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το είδος των καθηκών του, το προφίλ της δουλειάς που θα αναλάβει, το είδος των ευθυνών του. Και αναφέρω αυτό το θέμα, όχι βέβαια είναι πολιτικό το λειτουργήμα, το παραπέμπουμε στην Επιτροπή Διοντολογίας και γίνεται μια σύγκριση των νέων καθηκόντων και ευθυνών με τα καθήκοντα και τις ευθύνες που είχε κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Επιτρόπου. Αν λοιπόν υπάρχει μια δυνητική σύγκρουση συμφερόντων, η Επιτροπή Θετολογίας ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει τον, τον ενδιαφερόμενο πρώην Επίτροπο να μην αναλάβει τη νέα θέση. Το ίδιο συνέ... Αυτό συνέβη με τον πρώην Επίτροπο Μακρύβη και μία θέση σε τράπεζα. Τα θέματα της αιτιολόγησης ε, ή των πορισμάτων της ε, Επιτροπής Διατολογίας ε, σκεφτόμαστε να τα δημοσιοποιήσουμε ώστε να είναι όλα προσιτά και διαφανή και να γνωρίζει ο κόσμος πώς κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση η Επιτροπή Διατολογίας. Ό,τι αφορά το θέμα της ανεξαρτησίας των Επιτρόπων, υπάρχουν τρία στάδια εδώ. Καταρχήν πριν την ανάληψη των καθηκόντων. Έχουμε το θέμα της δήλωσης των συμφερόντων, Έχουμε το όλο ζήτημα του πολιτικού ελέγχου που υπόκεινται οι επίτροποι και επίσης υπάρχει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, ο έλεγχος του Πρόεδρου της Επιτροπής, ο έλεγχος από το κοινό. Είναι προς συμφέρον μας λοιπόν να αποφεύγουμε σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό δεν σημαίνει ότι με το που αναλαμβάνουμε τη θέση δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, γιατί εξακολουθούμε να είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε οποιαδήποτε δυνητική σύγκρουση συμφερόντων ακόμη και μετά την λήξη της ε, θητείας του Επιτρόπου. Και μάλιστα η υποχρέωση κανονικά ισχύει διοντολογικά μέχρι καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Γιατί υπάρχει και δυνατότητα ασφαλιστικών μέτρων όταν παραβιάζεται αυτός ο διοντολογικός κώδικας ε, και χρόνια μετά την απώλεια της ε, θέσης του Επιτρόπου. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το σύστημα ελέγχων να το αποσαφηνίσουμε και να το κάνουμε πιο προσιτό και πιο γνωστό. Ο κύριος Στάις είπε ότι είναι καλό σημείο φετηρία η πρόταση αυτή για τη συζήτηση. Συμφωνώ μαζί σας κύριε Στάις και ευελπιστώ ότι αυτή η γενική παρουσίαση που έγινε προφορικά θα αντικατοπτριστεί και στο τελικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι υπό επεξεργασία όπως σας είπα και οι δικέ σα συστάσει είναι ευπρόσδεκτε, γιατί μπορεί να μην είστε πιο δημοφιλή και αγαπητή Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά σίγουρα έχετε κύρο. Πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και μα ενδιαφέρει η υποστήριξη τη Επιτροπή σα για τον κώδικα δεντολογία των Επιτρόπων, έστω και ενό μεγάλου τμήματο του κώδικα δεντολογία, αν όχι του συνόλου του. Κύριε Γκάιερ. Και κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στο ζήτημα των μεταβατικών αποδοχών αμοιβών. Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά ε, νομικιστή στην απάντησή μου, αλλά θα πρέπει να είμαστε σχολαστικοί και ακριβείς. Αν εξετάσουμε το θέμα των μισθών και των μεταβατικών ε, αμοιβών, θα δείτε ότι ρυθμίζονται από ένα συγκεκριμένο άρθρο της συνθήκης που μιλά για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τους δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τους επιτρόπους. Και αυτή ήταν απόφαση του Συμβουλίου. Δεν υπάρχει δικαίωμα πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό που προσπαθούμε τώρα είναι να ενεργήσουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας και να αποσαφηνίσουμε τους κανόνες για τους επιτρόπους με τη μορφή του κώδικα δοντολογίας και να αποφύγουμε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων ή να αποφύγουμε πιθανή εμ, αντιδεντολογική συμπεριφορά επιτρόπων. Βέβαια, το θέμα των μεταβατικών αποδοχών είναι ένα θέμα που έχει προβληθεί ιδιαίτερα στον τύπο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ενδιαφέρει και το κοινό. Γι' αυτό και θα πρέπει να το εξετάσουμε ενδελεχώς. Πάντως, αρμόδιος για την απόφαση είναι το Συμβούλιο. Ο αρμόδιος φορέας. Εμείς θα το εξετάσουμε, θα το αναλύσουμε διεξοδικά, αλλά σε τελευταίο βαθμό την απόφαση τη λάβει το Συμβούλιο. Τώρα, πώς θα χειριστούμε το θέμα των εγγράφων. Μέχρι στιγμής ε, είπαμε ότι θα ενημερώνουμε, θα ενημερώσουμε το κείμενο του κώδικα διοντολογίας και αν οι αλλαγές που σας πρότεινα γίνουν δεκτέ και από του υπόλοιπους επιτρόπους, θα προσαρμόσουμε την απόφαση την απόφασή μα και για την Επιτροπή Διοντολογία. Αυτά θα είναι τα δύο έγγραφα, κώδικα διοντολογία και έγγραφα για την Επιτροπή Διοντολογία, που θα πρέπει να επικαιροποιηθούν αν θα ισχύσουν νέες, νέοι κανόνε διοντολογία. Τώρα, πώ θα αποτρέψουμε επιρροή των κρατών μελών στους επιτρόπους, πώς θα διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία των επιτρόπων και τον επηρέαστο από τα κράτη-μέλη. Ελπίζουμε ότι όλοι θα σεβαστούν τη συνθήκη, γιατί προβλέπει με σαφήνεια ότι οι επίτροποι θα πρέπει να είναι απολύτως ανεξάρτητοι, δεν μπορούν να δεχθούν ε, ή να επιδιώξουν συμβουλή καθοδήγηση από οποιαδήποτε οργάνωση ή από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αυτά τα λέει καθαρά και ξάστερα η συνθήκη που προβλέπει και την υποχρέωση των κρατών μελών να μην επιχειρήσουν να επηρεάσουν το έργο των επιτρόπων, αρκεί λοιπόν να τηρήσουμε τη συνθήκη. Επίσης έχουμε και τον επίσημο όρκο που δίνουν οι επίτροποι στο Λουξεμβούργο. Όλοι ε, οι επίτροποι που αναλαμβάνουν το καθήκοντά τους ορκίζονται ε, επίσημα ότι δεν πρόκειται να δεχτούν οδηγίες ή εντολές από οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε οργάνωση. Και πολύ συχνά, συμφωνώ μαζί σας, ασχολούμαστε με θέματα που είναι ακαθόδη για την πατρίδα μας, αλλά αυτό είναι θέμα δεοντολογίας, όχι μόνο για την Επιτροπή, αλλά και για τα κράτη-μέλη, που δεν πρέπει να προσπαθήσουν να επηρεάσουν κάποιον επίτροπο. Σε ό,τι αφορά τα γραφεία, τα προσωπικά γραφεία των επιτρόπων και το επιτελείο των συνεργατών τους. Μέχρι στιγμής είχαμε σαφείς κανόνες για τη σύνθεση του γραφείου του Επιτρόπου, όσο αφορά το μέγεθος, για το πόσα μέλη θα παρτίζετε, πόσους υπαλλήλου και θα πρέπει οι υπάλληλοι αυτοί να προέρχονται τουλάχιστον από τρεις χώρες. Δεν υπάρχουν δηλαδή γραφεία που να παρτίζονται μόνο από υπηκόους ενός κράτου. Θα πρέπει τουλάχιστον να προέρχονται από τρεις διαφορετικές χώρες ε, η βοήθεια του Επιτρόπου και να εξασφαλίσει φυσικά πνεύμα συνεργασίας, μια καλή ατμόσφαιρα και αυτό είναι σημαντικό να επικρατεί ένα κλίμα συνεργασίας στο γραφείο. Τώρα για, τις, για τους κανόνες σε ό,τι αφορά πόσα μέλη του γραφείου πρέπει να είναι μόνιμοι πάλι και πώς συμβασιούχοι και για το θέμα αυτό υπάρχουν κανόνες. Αυτή τη στιγμή πάντως προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε ότι αν υπάρχουν προθέσεις ε, για πρόσληψη συγγενούς ή συντρόφου ή συζύγου του Επιτρόπου στο γραφείο, αυτό πλέον θα είναι αδύνατο, θα αποκλείεται τέτοια πιθανότητα με βάση τη νέα πρόταση για το κώδικα δεντολογίας. Θέλουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε τέτοια δυνατότητα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε Σεφκόβιτ, για τις εισηγήσει σα και για τι απαντήσει που δώσατε. Σα ευχαριστούμε για την παρουσία σα εδώ και περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσης διάταξη, το σημείο 6. Passiamo al punto 6, la relazione speciale della Corte. Ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 4 του 2010 για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του καθεστώτος κινητικότητας του προγράμματος Λεωνάρντο Νταβίντσι και αν αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Δίνω το λόγο στον εισηγητή Πατριτσέλο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και τη κυρία Γκρέσλο που είναι η συντονίστριά μας που με βοήθησε να δουλέψω πάνω σε αυτό το θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είναι γνωστό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας το Μάρτιο του 2000 είχε ορίσει ως στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το να αποτελέσει μια οικονομία που θα βασίζεται στην γνώση μέχρι το 2010. Γνώση στην οποία προέρχεται από την παιδεία. Με βάση τα όσα αποφασίστηκαν στη Λισαβόνα, σε η διαδικασία της Κοπεχάγη που ξεκίνησε το 2002 από τους υπουργού ε, Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέσπιζε τον στόχο να ε, υπάρξει εθελοντική ε, επαγγελματική κατάρτιση για να προωθηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη αλλά και η αμοιβαία αναγνώριση των ε, πτυχίων ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα των εργαζομένων στην Ευρώπη. Στη συνέχεια η Κομισιόν ε, έκλεισε διάφορες ε, μάλλον συμπεριέλαβε μέσα στο πρόγραμμα διαβίου κατάρτισης που θεσπίστηκε το 2006 τέτοιου είδους προγράμματα για την προώθηση ανταλλαγών σε, σε τομείς που είναι νευραλική σημασία για την ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα στο πρόγραμμα για τη μόνιμη κατάρτιση συμπεριλαμβάνεται το υποπρόγραμμα Λεωνάρντο Ταβίντζη το οποίο προέκυψε με στόχο να εφαρμόσει την πολιτική κατάρτισης και επαγγελματική κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Leonardo του Νταβίντζη βασίζεται κυρίως σε προγράμματα κινητικότητας που αντιπροσωπεύουν το πιο σημαντικό κομμάτι του προγράμματος και επιτρέπουν σε οργανώσεις που λειτουργούν στον τομέα της παιδείας και της επαγγελματικής κατάρτισης να στείλουν τους συμμετέχοντες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να τους προσφέρει λοιπόν τη δυνατότητα να βελτιώσει τις ε, ικανότητές του, τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του. Επειδή πρόκειται λοιπόν για ένα πρόγραμμα για την οποία γενική ευθύνη έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που στους διάφορους ελέγχους εποπτείας της εφαρμογής του προγράμματος, σε συνεργασία με τις αρχές, τις εθνικές του κάθε, της κάθε χώρας, εφαρμόζει το πρόγραμμα. Με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα και ξέρω ότι είναι και ο δόκτωρ Ντέβισον που είναι σήμερα εδώ και διάβασα λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο ε, είχε στόχο να καθορίσει αν η διαχείριση του προγράμματος Λονάρντο, όπως έγινε από την Κομισιόν, επιτρέπει την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Η ανάλυση που έκανε ο κύριος Ντέβιτσον ε, δίνει ένα σαφές και λεπτομερές πλαίσιο της κατάστασης πρόοδου, δίνοντας χώρο για κάποιο προβληματισμό που θέλω να, σας, ε, να μοιραστώ μαζί σας. Καταρχήν, Ξεκινώντας από τα πορίσματα του ελέγχου του ελεγκτικού συνεδρίου, Συμμερίζομαι ότι η επεξεργασία και ε, η εφαρμογή του προγράμματος θα μπορούσε να δώσει αποτελέσματα απτά. Υπάρχουν όμως μια σειρά προβλήματα που ελπίζω μπορούν να αντιμετωπιστούν από την Κομισιόν όσο γίνεται νωρίτερα, ώστε ο προγραμματισμός να γίνει ακόμα πιο ικανοποιητικός και να ε, μπορέσει να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί. Ανάμεσα στα μεγαλύτερα προβλήματα πρέπει να διαπιστώσουμε ε, με τα μας ότι η Κομισιόν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να, να μετρήσει τα αποτελέσματα του προγράμματος λόγω ελλείψεων που υπάρχουν στο σύστημα παρουσίασης των ε, εκθέσεων που, των αναφορών που γίνονται αυτή τη στιγμή. Έχει γίνει η μελέτη για ένα γενικό σύστημα που θα έχει στόχο την αξιολόγηση και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος Λεωνάρδο και η Κομισιόν θα έχει τρία χρόνια Μάλλον, τρία χρόνια μετά την έναρξη του προγράμματος δεν μπορεί ακόμα να αξιολογήσει σε ποιο βαθμό επιτυγχάνονται οι προκαθορισμένοι στόχοι. Όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγηση των υποψηφίων και την επιλογή των προγραμμάτων των συμμετεχών των χωρών, πρόκειται για διαφανεί και καλά διοργανωμένε μεθόδου που συμφωνούν με τι διατάξεις της Κομισιόν. Όμως υπάρχουν ε, κάποιε αδυναμίες, όπως για παράδειγμα το γεγονό ότι οι υποψηφιότητε γίνονται δεκτές ακόμα κι αν η περιγραφή του περιεχομένου, του στόχου, του κόστους και των ε, αποτελεσμάτων δεν ήταν ε, επαρκής. Η επιπλέον ε, το πρόγραμμα δέχτηκε διάφορες επικρίσεις από συμμετέχοντες που, που σημείωσαν διάφορα προβλήματα όσον αφορά τους, τους εταίρους υποδοχής σε άλλες χώρες. Για διάφο, πολλούς και διάφορους λόγους. Καταρχήν δεν υπήρχαν ε, κατάλληλες γλωσσικές γνώσεις αλλά και υπάρχουν διάφορες πολιτιστικές ε, διαφορές. Γι' αυτό θα ήταν σκόπιμο η Κομισιόν να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τις πρόοδους που έχουν επιτευχθεί όσον αφορά την ε, προσπάθεια που φαίνεται να είναι απαραίτητη ώστε να υπάρχει ένα μέσο που θα μπορεί να λύσει τις, τα προβλήματα και τις δυσκολίες των υποψηφίων στην αναζήτηση εταίρων ή συνεργατών για την υποδοχή των ε, υποψηφίων στις άλλες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί το σύστημα πληροφορικής, να βελτιωθεί η στήριξη των συνεργατών υποδοχής, να αναπτυχθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης των ετοιμάτων για, πρόγραμμα, για προγράμματα, άρα τότε το πρόγραμμα θα είναι όντως επικοδομητικό για τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι επιδιώκουν τους στόχους για τους οποίους έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος ε, εδώ από την Κομισιόν που θέλει να παρέμβει ή από το ελεκτικό συνέδριο βέβαια. Κομισιόν κανείς. Μάλιστα παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ευπρόσδεκτη την έκθεση του Ευρωπαϊκού του Ελεγκτικού Συνεδρίου και χαίρεται για την ε, αγαστή συνεργασία και το θετικό συμπέρασμα της έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου σε ό,τι αφορά την ποιότητα και τη διαχείριση καθώς και τον έλεγχο του προγράμματος και το συμπέρασμα του Ελεκτικού Συνεδρίου ότι χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά το πρόγραμμα λειτουργεί αποτελεσματικά. Ας μην ξεχνούμε ότι ο έλεγχος κάλυπτε κυρίως ε, τα έτη 2007 και 2008, τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας δηλαδή του προγράμματος. Αυτό σε μεγάλο βαθμό εξηγεί και το συμπέρασμα του ελεκτικού συνεδρίου για πολλά και διάφορα σημεία του ελέγχου. την πρώτη διετία εφαρμογής όλα τα συστήματα διαχείρισης δεν είχαν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή και ήταν δύσκολο να καταμετρηθεί ο αντίκτυπος των πρώτων σχεδίων που είχαν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Da Vinci. Γιατί οι συνέπειες ε, φαίνονται χρόνια μετά την εφαρμογή. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε σε πολλές ε, εύστοχες παρατηρήσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου τα επόμενα χρόνια, μετά το 2008. Γι' αυτό και μπορούμε να δεχτούμε τα περισσότερα, τις περισσότερες συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου και μάλιστα ήδη έχουμε εφαρμόσει την πλειοψηφία αυτών των συστάσεων, είτε πλήρως είτε μερικώς. Μία από τις αδυναμίες που επισημαίνει η έκθεση είναι το γεγονός ότι οι δείκτες αντικτύπου δεν εγκρίθηκαν από την αρχή του προγράμματος παρά μόνο τρία χρόνια μετά την θέση σε ισχύ του προγράμματος. Και ε, υπήρχε στην αρχή διαφωνία ως προς την θέσπιση τέτοιων δικτών. Όντως, η διαδικασία θέσπισης δικτών ήταν αρκετά χρονοβόρα και δύσκολη εξαιτία της πληθώρας των στόχων που περιείχε η νομική βάση. Για να ληφθούν λοιπόν οι ε, υπόψη όλοι οι στόχοι και να θεσπιστούν δείκτες για, για αυτούς τους 60 στόχους ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Και μάλιστα από το δίδαγμα αυτό θα καθοδηγηθούμε και στο επόμενο πρόγραμμα. Είχαμε και την επιτροπή του προγράμματος και ήδη από του χρόνου θα έχουμε τα πρώτα δεδομένα από το σύστημα πληροφορικής ώστε να εξασφαλιστεί και η συνέχεια. Φυσικά δεν περιμέναμε την έκθεση αυτή για να καταλήξουμε σε ποσοτικούς δείκτες ό,τι αφορά την εφαρμογή του προγράμματος. Και πολύ γρήγορα ε, είμαστε σε θέση να πούμε πόσοι συμμετείχαν, τι κονδύλια δόθηκαν, ποιο ήταν το επίπεδο των επιδοτήσεων, ποιε ήταν οι κινήσεις, ε, η κινητικότητα μεταξύ των κρατών μελών. Όλες αυτές οι πληροφορίες ήταν ήδη στη διάθεσή μας από την αρχή και φυσικά συνεχίζουν να συλλέγονται και είναι πολύ σημαντικές. Έχουμε και ένα σύστημα feedback ε, των συμμετεχόντων ε, στο πρόγραμμα κινητικότητας του Λεωνάρντο ε, και έτσι έχουμε και την ποσοτική αξιολόγηση εκ μέρους των ίδιων των δικαιούχων του προγράμματος, των συμμετεχόντων. Κάτι που ήταν πολύ θετικό για την διοργάνωση του προγράμματος και την ανάλυση του αντικτύπου του στους ίδιους τους δικαιούχους. Ήδη από την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος είχαμε τέτοια σχόλια και feedback από τους ενδιαφερόμενους. Δυσκολία αντιμετωπίσαμε με μία σύσταση του ελεκτικού συνεδρίου που αφορούσε το ρόλο των εθνικών οργανισμών στις χώρες υποδοχής για την οργάνωση της υποδοχής των συμμετεχόντων. Γιατί το πρόγραμμα ποτέ δεν λειτουργήσε με τέτοιο τρόπο. Φυσικά οι οργανώσεις που στέλνουν μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν και την ποιότητα της φιλοξενίας και εμείς έχουμε και το feedback, τα σχόλια των συμμετεχόντων που τα αξιοποιούμε και νομίζω ότι θα ήταν υπέρμετρη η ευθύνη ε, στις ε, αρχές της χώρας υποδοχής για την ε, διοργάνωση της υποδοχής. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό άχθος αυτό για τις αρμόδιες αρχές της χώρας υποδοχής. Γι' αυτό και είχαμε πρόβλημα αυτή τη σύσταση. Σε ό,τι αφορά την αναζήτηση εταίρων, θα ήθελα να σας εξηγήσω ότι από την αρχή του προγράμματος είχαμε ε, μια τέτοια βάση δεδομένων αναζήτησης ε, εταίρων, αλλά χωρίς δυνατότητα εξασφάλισης της ποιότητας όλων των πληροφοριών της βάσης δεδομένων, χωρίς αξιόπιστες πληροφορίες, η βάση θα είχε μάλλον αρνητικό αντικτύπο παραθετικό. Και αυτή τη στιγμή διαρευνούμε νέες δυνατότητες σε ό,τι αφορά την έρευνα των εταίρων, γιατί όντως αυτό είναι ένα από τα κριτήρια επιτυχίας της εφαρμογής του Λεωνάρτο. Σας ευχαριστώ και με στη διάθεσή σας για να λύσω κάποιες απορίες αν έχετε. Σας ευχαριστώ, όπως το ελεκτικό συνεδρίο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους βουλευτές και της Επιτροπής σας που συμπεριέλαβαν το θέμα αυτό το σημαντικό αυτό θέμα στην ημερήσια διάταξη τη σημερινή. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον κύριο Πατριτσέλο για πολύ, το πολύ ισορροπημένο του έγγραφο εργασία. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Νομίζω ότι συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω επίσης για τα καλά λόγια σας. Ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πολλά καλά λόγια είπε για τη συνεργασία μας. Θα ήθελα να πω το ίδιο πιστεύουμε και εμείς. Ήταν εξαιρετική η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σε πολλά σημεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε τις συστάσεις και καλωσόρισε την εκθεσή μας. Κάποια σχόλια ίσως θα δικαιολογούσαν το ότι παίρνω το λόγο σήμερα. Πρώτου περάσω όμως αυτά. Να πω ότι σημείωσα πρόσφατα ότι στις 19 Οκτωβρίου ο Επίτροπος απέστειλε έγγραφο για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είδα κάποιες προτάσεις που είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Άρθρο 4, σελίδα 20 Χρειάζεται στοχευμένη εκχώρηση των κονδυλίων. Επίσης, στα συμπεράσματα αναφέρεται ότι ο αυριανός προϋπολογισμός θα πρέπει να έχει ως στόχος ε, πραγματικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων. Η έκθεση αυτή νομίζω ότι αυτά τα θέματα αφορά και αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι για παράδειγμα οι στόχοι αυτοί τους οποίους ε, αναφέρεται για παράδειγμα την βελτίωση της διαφάνειας και του καθεξής, θα πρέπει να διατυπωθούν με πιο ευφυή τρόπο. Αυτό πραγματεύεται η έκθεση. Για παράδειγμα, στο κεφάλαιο 40-48 ότι θα πρέπει να είναι εφικτό το πρόγραμμα και πραγματοποιήσιμο, το οποίο δεν ισχύει για το πρόγραμμα Λεωνάρντο, αλλά αν θυμάμαι καλά και στις 17 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να βελτιώσει τα στοιχεία αυτά, να διορθώσει αυτά τα κενά. Και ότι επίσης θα συμπεριληφθεί και το σύστημα IT και ότι αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί. Το μέλλον λοιπόν προδιαγράφεται λαμπρό για το πρόγραμμα Λεωνάρντο. Καλό είναι να ακούει κανείς καλά λόγια για την έκθεση, αλλά ακόμα καλύτερο είναι αν η έκθεση αυτή οδηγήσει σε ευφύ αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, να περάσουμε σε ένα άλλο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά την επίσκεψη της κοινή αντιπροσωπείας της Επιτροπής Προϋπολογισμού με την Επιτροπή Προϋπολογισμού στην Κροατία. Είχαμε την τελική έκθεση που έδινε ε, την αναφορά σε μια, για μια πολύ σημαντική επίσκεψη που κάναμε στην Κροατία. Σημαντική επίσκεψη διότι είναι μια χώρα η οποία σκοπεύει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα έπρεπε να κάνουμε μια αξιολόγηση της κατάστασης για πολύ λεπτά ζητήματα. Επιτύχαμε και μια συμφωνία για την έκθεση που και εγώ θεωρούσα πολύ καλή και δεν την ε, χρειάζεται να την αναφέρω πάλι γιατί την έχετε στους φακέλους σας. Εχθές ε, έλαβα μια επιστολή του συναδέλφου Deutsch που είπε ότι κατά την άποψή του έπρεπε κάπως να τροποποιηθεί η έκθεση αυτή ώστε να λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Κροατία στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Μάθαμε και ότι ο, επίτροπο, ο συνάδελφος Γκόραν της Επιτροπής Υπερπολογισμού συμφωνεί. Τώρα όμως δεν βλέπω τον συνάδελφο Ντόιτς. Θα μπορούσαμε ίσως να ζητήσουμε αυτή την συμβολή μέσω mail από πλευράς του συναδέλφου Ντόιτς να το δούμε με τους συναντονιστές και να δούμε αν συμφωνούμε για να ενταχθεί και αυτό το, αυτή η τροποποίηση και θα τροποποιήσουμε την έκθεση. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς να παρέμβει. Μία ερώτηση μόνο έχω να κάνω. Υπάρχει κάποια διαδικασία η οποία ακολουθείται για την έκθεση αυτή, γιατί όντως ο συντονιστή των, σοσιαλιστών, κύριο Φέρμ, συμμετείχε και στην αντιπροσωπεία, μου είπε ότι δεν συμφωνεί με την γενική νοτροπία που διέπει το έγγραφο του εισηγητή. Ίσως ε, επισερχόμαστε σε υπερβολικές ε, λεπτομέρειες. Αλλά σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κροατία δεν τα λαμβάνουμε σωστά υπόψη. Πώς θα ακολουθήσουμε λοιπόν τη διαδικασία, τι διαδικασία θα ακολουθηθεί. Θα προδίνουμε κάποιες συναλλακτικέ διατυπώσεις, κάποιες προσθήκες. Σε ποιον θα τις αποστείλουμε. Η κυρία Γκρέσλε διάβασα τις συστάσεις και το email του συναδέλφου ΦΕΜ και θεωρώ ότι οι πολιτικοί σε θέματα εξωτερικών θεωρούν ότι αν ρυθμίσουμε τα πάντα θα βελτιωθεί ο κόσμος γιατί η εμπειρία όμως είναι διαφορετική. Διάβασα τις συστάσεις, είναι σαφείς αλλά δεν είναι υπερβολικά αρνητικές και κοιτάζοντας τα συμπεράσματα του Λεκτικού Συνεδρίου του 2009 υπάρχουν προβλήματα στην Κροατία. Και στην ε, έκθεση αναφέρεται ότι τελικά συμφωνούν τα κράτη-μέλη. Κοιτάξτε, το τρένο θα προχωρήσει με την έκθεση αυτή και χωρίς την έκθεση αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας για να βελτιώσουμε, να διορθώσουμε τα προβλήματα. Υπάρχουν και κάποιες εκθέσεις πρωτοβουλίας σε ό,τι αφορά τα μέσα για τη διαδικασία, την προνταξιακή, θα συμπεριληφθεί και η Κροατία. Διάβασα την έκθεση, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο σαφής πια. Είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση όμω και η δική μου η εκτίμηση σε σχέση με του πολιτικού που ασχολούνται με τα εξωτερικά που, που είναι πάντα υπεραισιόδοξοι. Ήταν αρκετά σαφές και το email του κυρίου Φέρμ. Δεν ανέφερε τι θα πρέπει να αλλάξει συγκεκριμένα, απλά είχε μια γενική κριτική στάση. Εμείς θα μπορούσαμε να αποτεχτούμε το έκθεση όσο έχει. Κοιτάξτε, εγώ συμμετείχα σε αυτή την αντιπροσωπεία και θα πρέπει να σα πω τα τελικά αποτελέσματα που επιτύχαμε με αυτή την έκθεση ήταν σωστά. Επιπλέον, θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι τα σημαντικά θέματα της ε, ανεξαρτησίας του δικαστικού κατά πολέμηση της διαφθοράς δεδομένων των προβλημάτων που υπήρξαν στην Κροατία καλύτερα είναι να είμαστε λίγο πιο αυστηροί. Εγώ ειλικρινά σας λέω αφού έχει εγκριθεί από όλους ότι διατηρούσα για το μέλλον, ε, μετά από την πρόταση του Γκέιρ, εγώ θα έλεγα να υιοθετήσουμε το κανόνα που έχουμε υιοθετήσει μέχρι στιγμή. Ότι από τη στιγμή που υπάρχει συνένεση, ε, ε, κυκλοφορεί, μάλλον άμα υπάρχει συνένεση και μετά εγκρίνεται. Γιατί δεν χρειάζεται κάθε φορά να αρχόμαστε ξανά συζητάμε όλα τα θέματα. Ωραία λοιπόν, παύση 10 λεπτών τώρα, αφού έχουμε ψηφοφορία σημαντική στις 5, θα τα πούμε στις 5.